Ευχαριστώ λίγη η συζήτηση και αύριο 11.30 ώρα Πέμπτη ε, θα γίνει ψηφοφορία. Αύριο θα είναι η επόμενη συνεδρίαση 25 ε, Φεβρουαρίου από τις 9 και 30 ως τη 1. Η έκθεση έχει 9 μέχρι την 1. Ε, Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους τεχνικούς και τους διερμηνείς που βοήθησαν να ολοκληρώσουμε το βράδυ και σας ε, ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρία.